ξεκινήσουμε την συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Σημείο 1. Έγκριση της, ημε... της ημερήσιας διάταξης. Δεν υπάρχουν προτάσεις για αλλαγές του σχεδίου που λάβατε. Υπάρχουν αντιρρήσεις τώρα μήπως από πλευρά σας. Όχι. Οπότε εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Σημείο 2. Ανακοινώσει του Προέδρου. Να σας ενημερώσω ότι ότι στη συνεδρίαση της 9ης Οκτωβρίου οι συντονιστές όρισαν τον κύριο Καβαντά ως εισηγητή για την άρση της ασυλίας της κυρίας Ίγκεμπορ Γκρέσλε, την κυρία Ρέγνερ ως εισηγήτρια για την άρση ασυλίας του κυρίου Στίβ Μπριουά, τον κύριο Σβιεύκα ως εισηγητή για την πρόταση κανονισμού που θα αντικαταστήσει το παράρτημα Α του κανονισμού 2015 κάθετος 845 για τις διαδικασίες αφαιρεγγιότητας. Εμένα ως εισηγητή για την γνωμοδότηση επί της απαλλαγής 2016 για το Γενικό Προϋπολογισμό της Ένωσης, τμήμα του Δικαστηρίου, τον κύριο Χρυσόγονο ως εισηγητή για τη γνωμοδότηση της ε, εποπτείας του δημοσιονομικού συστήματος και τη θέσπιση ενός Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου, την κυρία Χάουταλα ως εισηγήτρια για τη γνωμοδότηση ε, για τον πλουραλισμό των μέσων μαζικής ενημέρωσης και την ελευθεροτυπία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, στην ίδια συνεδρίαση, οι συντονιστές αποφάσισαν να μην γνωμοδοτήσουν για την Επιτροπή ΠΕΤΗ σε σχέση με την αναφορά υπαριθμών 0178 κάθετος 2017 και ο πρόεδρος ενημέρωσε σχετικά την Επιτροπή ΠΕΤΗ. Επίσης, δεν θα γνωμοδοτήσουμε στην, για την Επιτροπή ΕΚΟΝ όσον αφορά τους κανονισμούς που τροποποιούν τους κανονισμούς για την ολοκληρωμένε τις ολοκληρωμένες δημοσιονομικές αγορές, χρηματοπιστωτικές αγορές, με συγχωρείτε. Επίσης, δεν θα χρηματοδοτήσουμε για... προς την Επιτροπή ίντα για τη θέσπιση πλαισίου για τον έλεγχο των ξένων άμεσων επενδύσεων στην Ένωση. Και τέλος, δεν θα γνωμοδοτήσουμε ούτε για την Επιτροπή Γυναικών για την ισότητα των φύλων στον τομέα των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ένωση. Οι συντονιστές ενέκριναν δε το πρόγραμμα των ακροάσεων της Επιτροπής Γιούρη για το πρώτο εξάμεινο του 2018 που έχει επίσης πια εγκριθεί και από το Προεδρείο του Κοινοβουλίου. Οι συντονιστές συμφώνησαν για τη σημασία της σωστής εφαρμογής των αρχών ασυλίας. Δεύτερον, η ομάδα εργασίας Γιούρι Αύκο για την εφαρμογή και ε, της Διοργανικής Συμφωνίας για την καλύτερη νομοθεσία ολοκλήρωσε τις εργασίες του ε, σήμερα και ενέκρινε τις εκθέσεις δραστηριοτήτων και, τους και οι ο κύριος Ρέο Κόρμπερ και εγώ ο ίδιος, έγιναμε τις ε, συστάσεις για το χρονοδιάγραμμα που θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε στην έγκριση της έκθεσης ίδιας πρωτοβουλίας Γιούρι Αύκο και η πρώτη ανταλλαγή απόψεων θα γίνει στις Επιτροπές Γιούρη και Αύκο στις 28 Νοεμβρίου. Αυτά για τις αποφάσεις των συντονιστών και οι δικές μου ανακοινώσεις. Ε, σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων. Εάν δεν λάβω αντιρρήσει ε, ή ενστάσεις μέχρι το πέρα αυτή τη συνεδρίασης, τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Δευτέρας Οκτωβρίου 2017 και 9 η και 10 η Οκτωβρίου 2017 θα θεωρηθεί ότι εγκρίνονται. Συνεχίζουμε με το σημείο υπαριθμών 4 εξέταση του σχεδίου σύστασης για την ολοκλήρωση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης της συνθήκης του Μαρακέσε για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα για ανθρώπους που είναι τυφλοί, έχουν δυσκολίες όραση ή δεν μπορούν να διαβάσουν. Και το λόγο δίνω στον κύριο Άντερσον που είναι ο εισηγητής. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε το πακέτο Μαρακές περιλαμβάνει οδηγία και κανονισμό και ολοκληρώθηκε η διαπραγματευσή του και υπογράφηκε από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 31 Σεπτεμβρίου τρέχοντος. Αυτό το, αυτή η δέσμη εφαρμόζει τη συνθήκη του Μαρακές στο, στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που προβλέπει την πρόσβαση των ανθρώπων με δυσκολίες όρασης στα έργα τα οποία ήδη είναι ε, ε έχουν ήδη εκδοθεί. Τώρα πρέπει να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας ε, στην σύναψη της συνθήκης του Μαρακές. Εγώ καλωσορίζω την απόφαση του Συμβουλίου για την ε, ολοκλήρωση αυτής της συνθήκης. Είναι ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την πλήρη εφαρμογή αυτής της πολύ σημαντικής νομοθεσίας. Γι' αυτό και συστήνω στο σχέδιο σύστασή μου να ε, εγκρίνουμε την ολοκλήρωση της συνθήκης του Μαρακές. Thank uh, uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, κανείς ε, θέλει να πάρει το λόγο για αυτό το θέμα? Doesn't seem to be, be the case. the Commission to... Η Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Thanks a lot. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Όμως η Επιτροπή θέλει να συγχαρεί τον εισηγητή κύριο Άντερσον και να εκφράσει την ικανοποίησή της για την πρόοδο σε αυτό το σημαντικό θέμα, την κύρωση της συνθήκης του Μαρα... Μαρακές. Όπως είπε ο εισηγητής, το Συμβούλιο ήδη έχει καταθέσει σχέδιο απόφασης και τώρα βλέπουμε ότι και το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να προχωρήσει στην συγκατάθεση. Η συνθήκη του Μαρακές αποτελεί εδώ και καιρό προτεραιότητα της Κομισιόν και ανέκαθεν ήμασταν ικανοποιημένοι από την υποστήριξη που λάβαμε ε, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, τα τελευταία χρόνια υπήρξαν κάποιες δυσκολίες λόγω ζητημάτων που δεν είχαν να κάνουν με την ουσία της συνθήκης, αλλά είχαν να κάνουν με τι διεθνεί αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό, αλλά από ό,τι φαίνεται μετά από την απόφαση του Δικαστηρίου και τις πρωτοβουλίες του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου για κύρωση, το θέμα είναι πια στο δρόμο προς επίλυση και θέλουμε να υποστηρίξουμε πλήρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να συγχαρούμε και πάλι τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο σε αυτό το θέμα. Όχι. Να πω μόνο ότι η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών, εάν δεν κάνω λάθος, είναι 24 Νοεμβρίου. Μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Ολοκληρώνουμε λοιπόν την εξέταση αυτού του θέματος. Επόμενο θέμα είναι το υπαριθμόν 5. Εξέταση συμβαστικών τροπολογιών για τη δικαιοδοσία, αναγνώριση και επιβολή αποφασεών σε θέματα γάμου και θέματα γονικής ευθύνης καθώς και για θέματα διεθνών απαγωγών παιδιών. Πρόκειται για μια νέα διατύπωση, recast, και θα δώσω το λόγο στο... Ε, ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Σβιέφκα, τον εισηγητή που δεν είναι εδώ. Ε, ε, κάπου έχει κολλήσει από το αεροδρόμιο. Έρχεται. Θα σας διαβάσω αυτά που μου έστειλε. Και τα διαβάζω εξ ονόματός του.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 Εν ώψη τη ψηφορία ε, που θα γίνει αύριο, ο εισηγητή ε, θέλει να ευχαριστήσει όλου του και εισηγητέ ε, και το προσωπικό για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε για αυτό το θέμα και για το ότι καταλήξαμε στα σημαντικότερα θέματα. Η, η συμβαστική αυτή πρόταση εστιάζεται σε τρία βασικά θέματα. Πρώτον, η, ακρόαση τη άποψη του παιδιού, διαμεσολάβηση και τοποθέτηση του παιδιού στο εξωτερικό. Στόχο είναι είναι να επιτύχουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για το παιδί σε μια περίπλοκη κατάσταση, ε, σε περιπτώσεις ε, όπου υπάρχει επιμέλεια του παιδιού και όπου έχει υπάρξει και απαγωγή του παιδιού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο επιθυμούν επικαιροποίηση και ανανέωση των διαπραγματεύσεων με τα κράτη-μέλη με την ελπίδα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επειδή ακριβώ βρίσκεται σε διαδικασία διαμεσολάβησης, το Συμβούλιο στο μέλλον θα λάβει υπόψη του τα αποτελέσματα των ε, διαπραγματεύσεων με την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων. Αυτά λέει ο εισηγητής ο κύριος Σβιεύσκα. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην πρόεδρο της ε, ομάδας εργασίας ε, της Συμφωνίας Brussels ε, Βρυξέλλες 2α για να μας ενημερώσει για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητά μέλη του Κοινοβουλίου και συνάδελφοι, είναι τιμή για μένα που με κάλεσε ο κύριος Σβεύσκα να σας παρουσιάσω σύντομα τις διαπραγματεύσεις, πώς έχουν εξελιχθεί οι διαπραγματεύσεις μέχρι τώρα με το Συμβούλιο για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα. Χάλιντο Κόιτ είναι το όνομά μου και είμαι πρόεδρος της ομάδας εργασίας Βρυξέλλες 2. Υπήρξα πρόεδρος της ομάδας Βρυξέλλες 2 κατά διάρκεια της Εσθονικής Προεδρίας. Τα γνωρίζετε, οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν τον 16 τον Ιούλιο κατά διάρκεια της ε, Προεδρίας της Σλοβακίας δημιουργήθηκε μια πολύ φιλική ε, ατμόσφαιρα, καλό κλίμα για τις ε, συζητήσεις μας και αυτό το κλίμα συνεχίστηκε και με την Προεδρία της Μάλτας και της Εστονίας. Εξετάσαμε το κείμενο, πρώτη ανάγνωση, Μάρτιος του 2017, η δεύτερη ανάγνωση μετά αυτής της Μάλτας αφορά στον στο πεδίο και στους ορισμούς και το δεύτερο κεφάλαιο, η δικαιοδοσία, επίσης ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2017 από την Προεδρία της Μάλτας. Μέχρι τώρα η Εστονική Προεδρία είχε 9,5 ημέρες ε, συνεδριάσεων της ομάδας εργασίας και προβλέπονται και κάποιες άλλες ημέρες συνεδριάσεων το Δεκέμβρη. Κατά τη διάρκεια αυτών των συνεδριάσεων είχαμε πολλές και σημαντικές συζητήσεις, παραδείγματος χάρη ε, το θέμα της κατάργησης ε, των προβλέψεων και ποσοστώσεων να υπάρχει και η ακρόση της άποψη του παιδιού, η σχέση ανάμεσα στις ρήτρε συνεργασίας που προβλέπονται σε αυτόν τον κανονισμό και τη σύμβαση της Χάγης του 1996 και επίσης διασυνοριακή τοποθέτηση του παιδιού μπορέσαμε τη δεύτερη ανάγνωση του τρίτου κεφαλαίου για την διεθνή απαγωγή παιδιού και το κεφάλαιο 4 για τη συνεργασία ανάμεσα σε αρμόδιες αρχές σε θέματα γονικής μέρημνας. Αυτά τα ολοκληρώσαμε και θα ξεκινήσουμε την δεύτερη εξέταση του κεφαλαίου 6 που αφορά τις γενικές ρήτρε. Αυτά θα γίνουν το Δεκέμβρη και ελπίζουμε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες μας το Δεκέμβρη γιατί πρόκειται για λίγα μόνο άρτρα. Ε, θέλουμε το θέμα να πάει στο Τζάι του Δεκεμβρίου για να ε, ολοκληρωθεί και το θέμα όλων των υπόλοιπων αποφάσεων που αφορούν στην εξέκουα να υπάρχει ε, η σωστή διαδικασία για την κήρυξη της εκτελεστότητας, την εξεκουατούρ. Έχουμε λοιπόν τρεις δυνατότητες ε, με βάση τη Συμφωνία Βρυξέλλες 1 Εκεί προβλέπεται και κάποια στοιχεία από την Συμφωνία Βρυξέλλης 2. Το τρίτο προτινόμενο μοντέλο είναι ο συνδυασμό των δύο, δηλαδή να βρούμε κάτι το οποίο πραγματικά θα βοηθάει στα κρατημέλη, γιατί αυτό είναι ένα θέμα επί το οποίο ε, χρειάζεται η ομοφωνία. Το σύστημα Βρυξέλλης 1 και η τρίτη επιλογή αφορούν όλες τις προκλήσεις ε, που ισχύουν. Η απαγωγή του παιδιού αφορά ένα μεικτό σύστημα το οποίο μοιάζει με αυτά που ισχύουν τώρα, ε, κυρίως στις ε, προνομιούχες περιπτώσεις, αλλά η Συμφωνία Βρυξέλλες 1 προβλέπει την κατάργηση της διαδικασίας κήρυξης της εκτελεστότητας για τις υπόλοιπες αποφάσεις. Ε, υπάρχει το δικαίωμα της άμυνας κυρίως στις περιπτώσεις όπου έχουμε προνομιούχα κατάσταση και αυτό σημαίνει την ε, αντιπαράθεση σε δύο διαφορετικά κράτη-μέλη. Το αποτέλεσμα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου θα ε, δρομολογήσει εξελίξεις για την Βουλγαρική Προεδρία, η οποία θα επιληφθεί της δεύτερης ε, εξέτασης του τέταρτου κεφαλαίου. Από τη συνάντησή μας με τον κύριο Σβέφκα και την ομάδα του στις 8 Νοεμβρίου καταλήξαμε στο ότι οι τροπολογίες που προτείνονται από το Κοινοβούλιο, οι συμβαστικές προτάσεις κατατέθηκαν στο πλαίσιο της αναδιατύπωσης. Ε, το Συμβούλιο χαιρετίζει αυτή την κίνηση και θεωρούμε ότι και τα τρία αυτά θέματα ε, σας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Η ακρόαση της άποψης του παιδιού, η διαμεσολάβηση και η διεθνής τοποθέτηση του παιδιού. Αυτά είναι τα τρία βασικά θέματα που μας ενδιαφέρουν. Η ακρόαση της άποψης του παιδιού, αυτό ε, ακούστηκε κατά διάρκεια της Μαλτέζικης Προεδρίας τον Ιούνιο και αποφασίστηκε ότι το άρθρο 20 θα πρέπει να διατηρηθεί, που σημαίνει ότι προβλέπεται οριζόντια υποχρέωση να εισακούεται η άποψη του παιδιού. Αναφέρθηκε βέβαια με σαφήνεια ότι ο τρόπος με τον οποίο θα ακούγεται η άποψη του παιδιού αυτό ε, είναι θέμα εθνικής νομοθεσίας. Εμείς θέλουμε ένα εντάφιο το οποίο λέει ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα περιβάλλον φιλικό προς το παιδί για να ακουστεί η άποψή του. Το κείμενο του άρθρου 20 βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο άρθρο 12 της Σύμβασης των ΗΠΑ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και στην σχετική νομολογία ε, του, Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Επίσης αποφασίσαμε να, ακούμε, να διαφυλάξουμε και την παραβίαση αυτού του δικαιώματο του παιδιού, αλλά μόνο στο βαθμό που η παραβίαση βασίζεται στο άρθρο 20 και όχι στους διάφορους εθνικούς κανόνες. Δηλαδή, ειδικά στο δικαίωμα του παιδιού να ακουστεί η άποψή του. Για τη διαμεσολάβηση έχουμε ένα ξεχωριστό άρθρο στο κεφάλαιο περιεπαγωγής παιδιών για να είναι πιο ορατό το όλο θέμα και για να παραμένει και υποχρέωση των κεντρικών αρχών να βοηθούν στη διευκόλυνση της διαμεσολάβησης σε άλλες περιπτώσεις γονικής μέρημνας. Βασικά αναφερόμετα στη διαμεσολάβηση ή σε άλλες μορφές ε, διευθέτησης ε, διενέξεων που έχουν άμεση σχέση με την οδηγία περί διαμεσολάβησης. Νομίζω ότι και εδώ θέλουμε να έχουμε ένα περισσότερο οριζόντιο άρθρο, οριζόντιας εφαρμογής για τη διαμεσολάβηση. Επειδή όμως ήδη υπάρχει η οδηγία περί διαμεσολάβησης, τα κρατη κρατη ότι κάτι τέτοιο δεν είναι απαραίτητο. Σας είπα όμω ότι εμεί προσπαθήσαμε να συμπεριλάβουμε όσο δυνατόν περισσότερα στοιχεία. Η διαμεσολάβηση είναι πιο ορατή και αυτό το πράξαμε με ένα ξεχωριστό άρθρο. Όσον αφορά τώρα την διασυνοριακή τοποθέτηση. Είχαμε πολλές συζητήσεις το Σεπτέμβρη για την τοποθέτηση, δηλαδή κατά πόσο η διαδικασία που θα ισχύει θα είναι διαφορετική σχετικά με το πού θα τοποθετηθεί το παιδί, αν θα πάει σε γονείς, σε θεσμούς ή σε ανάδοχες οικογένειες. Και επίσης και για το πόσο καιρό θα διαρκέσει η τοποθέτηση. Θα είναι μακροπρο... μακροχρόνια ή βραχίδια ε, καταλήξαμε στο ότι δεν μπορούν να δοθούν απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, γιατί κανείς από εμά δεν ήξερε πού τραβιέται η κόκκινη γραμμή ανάμεσα σε μέλος οικογένειας και ανάδοχη οικογένεια, επειδή υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί της οικογένειας. Και το ίδιο ισχύει και για την μακροχρόνια και την βραχίδια τοποθέτηση. Πότε γίνεται μια τοποθέτηση βραχίδια ή ε, μακροχρόνια. Γι' αυτό αποφασίσαμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε πάνω σε ένα σύστημα που θα καλύπτονται όλες οι τοποθετήσεις εξαιρουμένων των περιπτώσεων όπου το παιδί θα ε, τοποθετηθεί στους γονείς του που ζουν στο εξωτερικό. Συγκεκριμένα, ε, αν θέλετε, σε ένα γονέα, μητέρα ή πατέρα. Επίσης, θέλουμε να προσθεθεί ένα εντάφιο που να εξηγεί ότι ακόλουθες περιπτώσεις θα καλύπτονται και αυτές, δηλαδή ορισμός ε, κηδεμόνων, όπου δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, αλλά επειδή ο κυδεμόνα ζει σε άλλο κράτο από το παιδί, το παιδί θα πρέπει να αλλάξει τοποθέτηση, ακριβώ επειδή θα έχει οριστεί εντωμεταξύ κυδεμόνα. Προτείναμε να επιτρέπουμε στα κράτη-μέλη να προβαίνουν σε ρυθμίσεις μεταξύ τους με στόχο να διευκολύνεται η διαδικασία διαβουλεύσεων, αλλά παρόλα αυτά θα πρέπει να δούμε πώ θα εξελιχθεί το θέμα και θα δούμε και τι κείμενο θα διατυπωθεί στο μέλλον. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την αγαστή συνεργασία. Το Συμβούλιο προσβλέπει στο να λάβει την έκθεση από το Κοινοβούλιο για τη Συμφωνία Βρυξέλλες 2α για τον κανονισμό Βρυξέλλες 2α. Και αν θέλετε και η ε, μελλοντική Προεδρία θα σας ενημερώσει για το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και βεβαίως αν έχετε ερωτήσεις είμαι στη διάθεσή σας. Now, uh, the, the... Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν κάποια μέλη θα ήθελαν, κάποιοι βουλευτές θέλουν να κάνουν σχόλια και ω Μπούντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εκπρόσωπο του Συμβουλίου για αυτές τις εξηγήσεις. Και να ευχαριστήσω και τον κύριο Σβιέτσκα για τις προσπάθειες του. Η έκθεση αυτή είναι ιδιαίτερα ε, λεπτή, διότι μιλούμε για ανήλικους και για την προστασία τους, καθώς επίσης και για το πώς θα πρέπει να χειριστούμε ζητήματα σχετικά με αυτούς και ζητήματα αρκετά ε, λεπτά. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω την εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Είναι σαφές ότι αυτή η διαδικασία είναι δύσκολο να εφαρμοστεί. Για παράδειγμα, σε ορισμένε περιπτώσεις ένα κράτος μέλος λαμβάνει μια απόφαση ε, ενώ η ίδια απόφαση δεν θα έχει σε ένα άλλο κράτος μέλος. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Για παράδειγμα, λαμβάνεται απόφαση στην Ισπανία και το παιδί βρίσκεται στη Ρουμανία πώς θα μεταφερθεί αυτό το παιδί από το ένα κράτος μέλος σε άλλο, στο άλλο. Το βλέπουμε και στην πράξη ότι δεν επιτυχάνεται πάντοτε η εκτέλεση των αποφάσεων, των δικαστικών αποφάσεων αυτού του τύπου. Επίσης υπάρχουν ορισμένε χώρες όπως η Ρουμανία όπου υφίσταται ε, η η δυνατότητα σε περίπτωση διαζυγίου, αν συμφωνήσουν τα μέρη, οι ρυθμίσεις να γίνουν με τρόπο, ε, με φιλικό διακανονισμό ενώπιον ενός υπαλλήλου, κρατικού υπαλλήλου, όχι δικαστικού. Ε, υπάρχει και αυτή η διαδικασία. Μπορούμε να συνεχίσουμε, θα μπορούσε να συνεχιστεί αυτή η διαδικασία στο μέλλον. Πρόκειται για ένα, μια διαδικασία η οποία πραγματικά ωφελεί και τα δύο μέρη διότι ρυθμίζει διαφορές χωρίς εντάσεις. Επιπλέον μειώνεται ο φόρτος των ε, ε, δικαστηρίων. Πώς μπορεί επίσης να ε, μετακινηθεί ένας ανήλικος με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχουν άλλοι βουλευτές που θέλουν το λόγο, να ζητήσω από την εκπρόσωπο της Προεδρίας να απαντήσει την ερώτηση του κ. Μπούντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ελπίζω να κατάλαβα την ερώτηση. Πώς μπορεί να μεταφερθεί ένα παιδί από ένα κράτος σε ένα άλλο. Πρώτον, ε, προφανώς έχουμε την διαδικασία αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων. Η κατάρριξη του εξεκουάτουρ του, θα, γίνει, θα εγκριθεί από το Συμβούλιο το Δεκέμβριο. Θα σας πω τότε λοιπόν πώς ε, θα γίνεται πρακτικά ε, η δήλωση του εκτελεστού. Ε, όμως το Συμβούλιο έκανε αυτό που έπρεπε ως τώρα, δηλαδή προσπάθησε να καταστήσει πιο ευρείε τι αρμοδιότητε τη κεντρική διοίκηση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε διάφορες, διαφορετικά σενάρια. Υπάρχει πλέον ο Κανόνα της ε, συνδρομής στην εφαρμογή δικαστικής απόφασης. Ε, όταν δηλαδή δεν εκτελείται με δεσμευτικά μέσα, υποχρεωτικά μέσα, ε, αλλά στην, όπως στην περίπτωσή σας προκύπτει ότι ένα παιδί θα πρέπει να μεταφερθεί σε ένα κράτος μέλος, οι κεντρικές αρχές μπορούν να συνδράμουν έτσι ώστε να βρεθεί ο τρόπος να γίνει είτε για παράδειγμα με, μέσω ενός ε, λειτουργού ο οποίος πηγαίνει να πάρει το παιδί σε άλλη χώρα ή συναντώνται στα σύνορα ή τέλος πάντων θα βρεθούν ad hoc ε, ε τρόποι για να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση. Αυτή είναι η απάντησή μου. Okay. Ε, ο κ. Σομπούντα ε, δείχνει ικανοποιημένος. Η κ. Äh, σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα σας ζητώ συγγνώμη να με δικαιολογήσετε που καθυστέρησα, αλλά ξέρετε καθυστέρησε το αεροπλάνο μου. Και στην ίδια πτήση ήταν και ο κύριος Σέπκεβια. Και γι' αυτό δεν έχει έρθει ακόμα. Βέβαια εγώ ήρθα νωρίτερα από εκείνον, ήμουν πιο γρήγορη. Εγώ λοιπόν είμαι η Σκιώδης εισηγήτρια εκ μέρους των σοσιαλιστών και θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε με τον κύριο Σιέσκα. Ε, υπάρχει μόνο ένα θέμα ε, που πραγματικά για μένα είναι κρίμα. Πρόκειται για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναδιατύπωση και εκεί προβλέπεται μόνο ο απαρχαιωμένος και πεπαλαιωμένος γάμος που υπάρχει εδώ και 100 χρόνια. Ότι αυτός, αυτή η μορφή γάμου λαμβάνεται υπόψη, αλλά όχι οι νέες μορφές συμβίωσης που υπάρχουν στα κράτη-μέλη. Έχω λοιπόν καταθέσει τροπολογίες και ξέρω κύριε Πρόεδρε, ε, θα πείτε ότι επειδή πρόκειται για recast, για αναδιατύπωση, αυτές οι τροπολογίες καταπίπτουν. Όμως για μένα είναι πολύ σημαντικό να καταστήσουμε σαφές ότι σήμερα υπάρχουν ε, πάρα πολλοί γάμοι που είναι πλέον ε, με τη μορφή ε, συμβίωσης. Υπάρχουν διάφοροι συνδυασμοί με παιδιά που δεν καλύπτονται από αυτή την νομοθεσία. Ε, θα ήταν λοιπόν σκόπιμο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο μέλλον να σκεφτεί ε, το πώς ακριβώς μπορούν να αντιμετωπιστούν και αυτοί οι συνδυασμοί. Διότι ε, αυτό που ενδιαφέρει πάνω απ' όλα είναι βεβαίως το καλό του παιδιού και σε τελική ανάλυση είναι αδιάφορο αν οι άνθρωποι είναι παντρεμένοι ή όχι. Αν είναι του ίδιου φίλου ή όχι. Αυτά δεν παίζουν κανένα ρόλο. Εφόσον ε, υπάρχει σχετική νομοθεσία που επιτρέπει τέτοιου είδους ε, συμβιώσεις, νομίζω ότι και αυτές θα πρέπει να καλύπτονται από την νομοθεσία. Γι' αυτό λοιπόν εκφράζω την παράκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα αυτά στο μέλλον να τα λάβει υπόψη. Δεν θέλω τώρα να αρχίσω να τσακώνομαι. Εγώ θέλω να ψηφιστούν αυτές οι τροπολογίες, αλλά σας λέω ειλικρινά, αυτό που επισημαίνω είναι απαραίτητο. Αυτό που βρίσκω πολύ καλό είναι οι συμβαστικές προτάσεις, στις οποίες κατέληξαν το καλό του παιδιού, το να ακούγεται η άποψη του παιδιού, Επίσης ε, τα παιδιά ανάλογα βέβαια με την ε, ηλικία τους, ε, στην ηλικία τους να προσαρμόζεται η όλη κατάσταση με βάση αυτή την ηλικία να προτείνεται ενδεχομένως η διαμεσολάβηση από το δικαστή και επίσης ε, θα μπορούσε και το κράτος σε κάποιες περιπτώσεις να επέμβει διότι σε τελική ανάλυση αυτό που ενδιαφέρει είναι όπως σας είπα το καλό του παιδιού η νομοθεσία να έχει κατά κύριο λόγο ο στόχο το καλό του παιδιού και όχι τους γονείς ή τους ε, συντρόφους ε, νομίζω ότι αυτές είναι καινοτομίε, είναι σημαντικέ εξελίξει και θέλω να ελπίζω ότι το Συμβούλιο θα δεχτεί να στηρίξει αυτέ τι εξελίξει. Thank you very much. Uh, I think that if Mr. Zwiefka would be here, I can guess that... Ε, νομίζω ότι ο κ. Ζιεύκα θα ήταν εδώ και θα απαντούσε ο ίδιος στο πρώτο κόμμα της παρέμβασής σας και ε, είμαι σίγουρος θα έλεγε ότι χαίρεται πως η Κομισιόν περιορίστηκε στο πεδίο ε, της αναδιατύπωσης, αλλά θα δώσω το λόγο και στην ίδια την Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε το λόγο. Και εγώ και, ο συνάλφος, η συνάλφος μου θα ήθελα να κάνω το εξή σχόλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά την Επιτροπή σας για την ε, συνεργασία που έδειξε τα, τους τελευταίους μήνες. Η συμβαστικέ τροπολογίες ε, τις οποίες ε, συζητούμε είναι ιδιαίτερα καλέ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ζιδιεύκα, ιδιαίτερο, που δεν, παρόλο που δεν είναι παρόν σήμερα, για, την, ε, για τον πολύ αποτελεσματικό τρόπο με τον οποίο συνεργάστηκε μαζί μα. Ακούσαμε από την Προεδρία ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση στο Συμβούλιο. Δεν υπάρχει λόγο λοιπόν να επαναλάβω τίποτα από αυτά. Θα ήθελα όμω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο για το γεγονό ότι εστιάζει τι τροπολογίε του σε θέματα που είναι πραγματικά σημαντικά σε αυτή την πρόταση αναδιατύπωση. Θεωρούμε το θέμα τη ακρόση του παιδιού, καθώ επίση και τη διαμεσολάβηση και τη διασυνορική τοποθέτηση των παιδιών είναι σημαντικότατε τροπολογίε. Ελπίζω ότι θα ολοκληρώσουμε αυτέ τι διαπραγματεύσει και για αυτά τα τρία ζητήματα με επιτυχία. Θα ήθελα να σχολιάσω με δύο λόγια την ε, ερώτηση της ε, κυρίας Γκέπχαρντ σε ό,τι αφορά την σχέση ανάμεσα στο παιδί και τους γονείς του οι οποίοι μπορούν να έχουν παντρευτεί με τον παραδοσιακό τρόπο ή με αστικό τρόπο. Θα σας πω πώς εφαρμόζεται σε αυτή τη στιγμή. Πράγματι, όταν η Κομισιόν υπέβαλε αυτή την πρόταση είχαμε συμπεριλάβει τουλάχιστον τον κανόνα της δυνατότητας οι γονείς να επιλέξουν το δικαστήριο για το διαζύγιο τους. Αυτό είναι δυνατόν για θέματα γονικής ευθύνης και πιστεύαμε ότι θα είναι ακόμα πιο χρήσιμο για θέματα διαζυγίου ή λύση του γάμου. Ε, η Κομισιόν όμως θα πρέπει πάντοτε να υποβάλει ε, αποδείξεις για το ότι το, κείμενο, ε, το προηγούμενο κείμενο είχε δημιουργήσει ε, προβλήματα. Δυστυχώς όμως σε αυτό το κομμάτι της πρότασής μας δεν καταφέραμε να αποδείξουμε ότι πράγματι ήταν προβληματικό το κείμενο. Γιατί πράγματι σύμφωνα με τον κανονισμό υφίστανται ε, κεντρικές αρχές που στηρίζουν τους γονείς σε ό,τι αφορά διαφορές για τα παιδιά τους σε διασυνορικές υποθέσεις. Αλλά δεν υπάρχουν τέτοιου είδους ε, ε, κεντρικές αρχές για γαμικές διαφορές. Δεν υπάρχουν στατιστικά και δεν υπάρχουν δεδομένα δεδομένα για να ε, ισχυριστούμε κάτι τέτοιο. Συνεπώ δεν θα πρέπει να σας εκπλήξει αν σας πω ότι μία εβδομάδα μετά την αποτυχία να περάσουμε ε, τη συμπεριληψή αυτού του θέματος ε, δεν, πάψαμε να είμαστε λυπημένοι διότι μία εβδομάδα μετά έγινε η ψηφοφορία στο Συμβούλιο για το θέμα του κανονισμού περιουσίας και έτσι ε, ξαναείδαμε την προσέγγιση μας για το γαμικό κομμάτι της πρόταση αυτής. Ε, όπως ξέρετε, ότι, όπως σας είπε και συνάδελφος, πρόκειται για θέμα το οποίο θα ψηφιστεί με ομοφωνία μόνο, οπότε ξέρουμε ότι δεν θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε ομοφωνία για οποιαδήποτε πρόταση έχει σχέση με την λύση ε, ε σχέσεις ε, ε, γονέων του ιδίου φίλου. Προκειμένου λοιπόν να μην θέσουμε σε κίνδυνο το κομμάτι που αφορά τα παιδιά, ε, αποφασίσαμε να μην συμπεριλάβουμε τις ε, να μην επιμείνουμε στις ε, προτάσεις μας για το θέμα της λύσης της σχέσης της οικογενειακής δηλαδή του οικογενειακού κομματιού του, της προτασής μας έτσι κι αλλιώς ε, νομίζουμε ότι ε, το θέμα των, για το θέμα των παιδιών το, το ζήτημα αυτό καλύπτεται και περιλαμβάνονται όλα τα ζευγάρια ανεξάρτητα του ίδιου φύλου διαφορετικού. Η νομοθεσία δυστυχώς πολύ συχνά ιστερεί έναντι της πραγματικότητας σε ό,τι αφορά την εξέλιξή της. Αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχουμε εξασφαλίσει αυτή την επιτυχία. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι τώρα εξαντλήσαμε το θέμα. Οπότε, μπορούμε να περάσουμε στην εξέταση δύο θεμάτων 6 και 7. Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης για τον κανονισμό που εισάγει μία ηλεκτρονική κάρτα ευρωπαϊκών υπηρεσιών συγγήτρια είναι η κυρία Γκέπχαρτ, στην οποία και δίνω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αυτές οι δύο προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή οδηγία και κανονισμός, αυτά ε, θέλουν να εισάγουν μια ηλεκτρονική κάρτα, όπου βέβαια ο όρος ηλεκτρονική κάρτα, e-card, δεν είναι ακριβής, γιατί αν δει κανείς τι προτείνεται, δεν είναι ακριβώς ηλεκτρονική κάρτα. Μπα περιπτώσει, σε δύο συναντήσεις ε, με σκιώδεις ηγητές ε, που είχα με τους ε, εισηγητές των διαφόρων πολιτικών ομάδων, συζητήσαμε διεξοδικά επί του θέματος και διατυπώσαμε και κάποιες ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή, ποια θα είναι η πραγματική προσθέμενη η αξία της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχοντας κατά νου και τα διάφορα εργαλεία τα οποία ήδη υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραδείγματο χάρη είναι ενιαίοι ε, συνομιλητές της οδηγίας ε, περί παροχής υπηρεσιών ή ε, επαγγελματική κάρτα, αμοιβαία αναγνώριση επαγγελματικών πτυχίων. Υπάρχουν δηλαδή συστήματα που βοηθούν οποτεδήποτε εμφανίζονται προβλήματα στα κράτη-μέλη. Υπάρχει ένα σύστημα που προβλέπει τη συνεργασία των ε, διοικήσεων ε, στα κράτη-μέλη. Αυτή τη στιγμή λοιπόν συζητάμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την ε, ψηφιακή πύλη, το Digital Gateway. θα ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει τελικά υπάρχουν αυτά τα εργαλεία και αυτή η ηλεκτρονική κάρτα τι θα προσφέρει παραπάνω, ποια θα είναι η προστιθέμενη αξία της, τι δεν υπάρχει με τα προηγούμενα εργαλεία. Οι απαντήσεις που έλαβα δεν είναι ικανοποιητικέ, διότι τελικά δεν καταλαβαίνω. Σας είπα ποια θα είναι η προστιθέμενη αξία με αυτή την ηλεκτρονική κάρτα. Βλέπω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που είναι τώρα παρούσα, ήταν παρούσα και στις τελευταίες συνεδριάσεις, τη στόχο ήδη πει ότι δεν είμαι ικανοποιημένη με τις απαντήσεις που μας έχει δώσει και δεν είμαι και ικανοποιημένη με τις απαντήσεις που δόθηκαν στην πολύ σωστή ερώτηση του κυρίου Μπούντα σχετικά με το κόστος που θα προκύψει αν υλοποιηθούν οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Άρα δηλαδή υπάρχουν αρκετά ερωτηματικά. Επειδή βέβαια πρέπει να ή έπρεπε να τοποθετηθώ για το λόγο αυτό έχω προετοιμάσει μία σειρά τροπολογιών. Πήγα σε μια δημόσια εκδήλωση με άμεσα ενδιαφερόμενους, όπου ήταν παρόν και ένας εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και ο Εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε σε αυτή την ε, εκδήλωση ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το κείμενο δεν είναι καλό, δεν είναι ικανοποιητικό και εκεί ε, είπα, ξέρετε φτάνει μέχρι εδώ. Σε τελική ανάλυση δεν είναι δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να βελτιώνει τα κείμενα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να στείλετε πίσω το κείμενο στην Επιτροπή και να μας στείλει πλέον, να μας υποβάλει πλέον η Επιτροπή ένα σωστό αιτιολογημένο κείμενο. Γιατί αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει να συσταθούν κάποιοι θεσμοί ή κάποιοι οργανισμοί στα κράτη-μέλη που θα είναι συνομιλητές ας πούμε του Solvit ή άλλων φορέων θα έλεγα α, εντάξει πράγματι προκύπτει προστιθέμενη αξία, προκύπτει τεχνογνωσία αλλά δεν προτείνεται αυτό αυτό που προτείνεται είναι κάτι το οποίο έτσι και αλλιώ έχουμε στην οδηγία περί υπηρεσιών και, και την οδηγία αυτή τι ε, την τονίσαμε τότε σε αυτή την οδηγία ότι δεν μας ενδιαφέρει η αρχή της καταγωγής αλλά η αρχή της ε, χώρας ε, διαμονής. Υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες ερωτήσεις πολλά ερωτηματικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι ε, κυρίως στον κατασκευαστικό τομέα είναι απαραίτητο να υπάρχει αυτή η ηλεκτρονική κάρτα. Εστιάζει δηλαδή η Επιτροπή στον κατασκευαστικό τομέα. Αλλά ξέρετε, αν υπάρχει ένα επάγγελμα που είναι διασυνοριακό, ε, είναι ακριβώς το ή τα επαγγέλματα στον τομέα των κατασκευών. Ως εκ τούτου θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και ένα θέμα που είναι σημαντικό και δεν έχει επιληθεί και δεν θα επιληθεί και με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι το θέμα της ασφάλειας. Αν δηλαδή θέλετε να κάνετε κάτι πραγματικά λογικό, τότε να ασχοληθείτε με τα προβλήματα που υπάρχουν και όχι να δημιουργήσετε ένα εργαλείο το οποίο στη τελική ανάλυση δεν προσφέρει τίποτα. Ε, και σκέφτομαι ότι αν κάνουμε αυτό που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή έχει καταθέσει δύο συγκεκριμένες προτάσεις. Αν τα κάνουμε όλα αυτά, ξαφνικά θα έχουμε μία ολόκληρη σειρά επικεδευματιών στα κράτη-μέλη, οι οποίοι θα έχουν κατοχήρωση στη χώρα τους, θα έχουν την ηλεκτρονική κάρτα, όμως οι άνθρωποι αυτοί δεν θα είναι επιτιδευματίες, θα είναι κατ' ουσίαν υπάλληλοι οι οποίοι θα έχουν αποσταλεί και παρόλα αυτά θα έχουν αποσπαστεί σε άλλο κράτος μέλος και παρόλα αυτά δεν θα καλύπτονται από τη σχετική οδηγία. Εγώ κάτι τέτοιο το θεωρώ απαράδεκτο. Παραδείγματο χάρη, στην περίπτωση αυτή με το κρέας, όταν η Ολλανδία ε, μήνυσε τη Γερμανία, το έπραξε ακριβώς επειδή υπάρχουν τέτοιου συστήματα και τότε είχαμε πει αυτό δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στα κοινωνικά συστήματα των κρατών μελών αντί να υπάρχει θεμητός ανταγωνισμός ανάμεσα στις επιχειρήσεις, στα κράτη-μέλη. Γιατί σε τελική ανάλυση όλοι τη θέλουμε την κοινή αγορά, αλλά να έχουμε κοινή αγορά υψηλού επίπεδου. Γι' αυτό λοιπόν εγώ αποφάσισα τις ε, τροπολογίες που τελικά είχα προτιμάσει να μην τις καταθέσω, αλλά να προτείνω να καταθέσουμε σύσταση στην καθήλια αρμόδια επιτροπή και αυτή η επιτροπή να απευθυνθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τη στείλει πίσω την πρότασή της. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Αυτό είναι το πιο λογικό που έχω να προτείνω. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο. Da, domnule președinte. Intervin în calitate de raportor din uh, umbră Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπούντα. Καταρχάς θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια που προσπάθησε πραγματικά να αποσαφηνίσει την πρόταση της Κομισιόν. Όμως πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Τα έγγραφα αυτά, η οδηγία και ο κανονισμός δηλαδή, θα πρέπει να βελτιωθούν κατά πολύ. Μπορούμε να απορρίψουμε βέβαια, μπορούμε να αρνηθούμε τελείως ε, αυτά τα κείμενα. Η μόνη επιλογή που έχουμε κατά τη γνώμη μας όμως δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ίσως να πρέπει να δούμε ποιες είναι οι δυνατότητες για βελτίωση. Γνωρίζουμε ότι όλοι έχουμε θέσεις πολύ διαφορετικές. Μπορούμε να δώσουμε μια προστεθέμενη αξία στην πρόταση της Επιτροπής. Πρέπει να έχουμε την προοπτική της ε, σαφήνειας. Τι συμβαίνει στην πράξη. Με αυτή την ηλεκτρονική ευρωπαϊκή ηλεκτρονική κάρτα που θα πρέπει να διευκολύνει κάποιες ε, διοικητικές διαδικασίες, θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει ένα να, να λειτουργήσει ως ένα μέσο στη διάθεση των πολιτών που να βελτιώσει την ζωή στα κράτη-μέλη. Πρόκειται για μια κάρτα που μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί εθελοντικά και αυτό θέλω να το τονίσω, δεν είναι υποχρεωτική. Άρα θα έπρεπε να κάνουμε μία πρόταση, ώστε ο πάροχος, ένας φορέας, ένας πάροχος, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ή να μην χρησιμοποιήσει την κάρτα αυτή. Κάτι άλλο σημαντικό είναι ότι ο πάροχος της υπηρεσίας θα πρέπει να μπορεί να κατανοήσει τι περιμένει ένα, κράτο, ένα κράτος μέλος. Βεβαίως υπάρχουν συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα τα οποία δεν αντιστοιχούν ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Για μας ο αρχιτέκτονας είναι διαφορετικός στο Ρουμανία από ότι ένας αρχιτέκτονας που εργάζεται στην Δανία. Θα έπρεπε δηλαδή να υπάρξει εναρμόνιση και σε αυτό το επίπεδο. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι η λύση πέρα από την απόρριψη. Και έπειτα υπάρχει και θέμα κόστους αν το κόστος είναι περιορισμένο και σας θυμίζω ότι το έχουμε ήδη συζητήσει στο Στρασβούργο αυτό το σημείο και είχαμε ακούσει τα όσα είχε να μας πει η Κομισιόν η απάντηση της Κομισιόν την περιμέναμε και γραπτός Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε λοιπόν περισσότερες πληροφορίες, όμως θα πρέπει να δούμε εάν θα λάβουμε αποφάσεις, αν μετά αυτές οι αποφάσεις θα τηρηθούν ή όχι. Κάτι άλλο που εγώ κάπως μελέτησα αυτό το θέμα, η οδηγία αυτή, αν τη συγκρίνουμε με αυτή για τις υπηρεσίες, μπορούν να συνεπάρξουν αυτές οι δύο οι τροπολογίε που εμείς θα υποβάλλουμε για αυτέ τι δύο εκθέσεις θα μας βοηθήσουν να σώσουμε αυτό το κείμενο γιατί επαναλαμβάνω πρέπει να δημιουργηθεί ένα μέσο το οποίο θα είναι προαιρετικό, δεν θα είναι υποχρεωτικό θα πρέπει ε, ο πάροχος της υπηρεσίας να επιλέγει αν θα το χρησιμοποιήσει ή όχι, να το βοηθήσει, να του διευκολύνει όμως να παραμένει επιλογή. Επιμένω λοιπόν γι' αυτό Ας κάνουμε τροπολογίες, ας δώσουμε μια προστιθέμενη αξία σε αυτήν την δυνατότητα και ας ελπίσουμε ότι εντωμεταξύ η Κομισιόν θα μας απαντήσει γιατί μέχρι στιγμή δεν μας την έδωσε γραπτό στην απάντηση. Uh, thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, η κυρία Merci, Monsieur le Président. Euh, je vous remercie de me laisser intervenir. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ποια είναι η διαδικασία συγκεκριμένα. Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που οφείλει μετά από αίτημα της κυρίας Γεύχαρτ και των σκιωδών να εξηγήσει τη θέση της επί της οδηγίας και να μας πει ε, σε τι αποτελεί απλοποίηση του δικαίου της Ένωσης. Η Κομισιόν προτείνει λοιπόν την, σύνταξη ενός κειμένου που λέει ότι μια επιχείρηση που ασκεί ασκεί νομίμως δραστηριότητες στη χώρα παρέλευσής του ή ο σεβασμός της ιδιαιτερότητας αυτών των χωρών, αυτής της συγκεκριμένη χώρας μπορεί να της δώσει τη δυνατότητα να κάνει μια παροχή στη χώρα όπου έχει ζητήσει αυτή την e-card. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει υπόψη την ελεύθερη κυκλοφορία και υπηρεσιών και θέλει έτσι να αφαιρέσει τον επιβολικό διοικητικό φόρτο. Όμως στην πράξη δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Επικρατεί πλήρης αοριστία για αυτή την πρόταση σε όλα τα επίπεδα δεν οδηγεί τίποτα σε απλοποίηση της νομοθεσίας και των ε, πρακτικών που επικρατούν και η κυρία Γκέπχαρτ πολύ σωστά μας το θύμισε ότι υπάρχουν ένα σωρό ευρωπαϊκά κείμενα για το θέμα της προστασίας του καταναλωτή, διγεία υπηρεσιών, αλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στις ε, διοικήσεις, στους διοικητικούς μηχανισμούς. Γιατί λοιπόν ακόμα ένα κείμενο, νέο κείμενο και αυτό είναι το ερώτημα της, της ε, εισηγήτριάς μας, ποια είναι η προστιθέμενη αξία αυτού του κειμένου και εγώ συμφωνώ απόλυτα με τη δική της γνώμη και με την ανάλυση που έκανε. Ε, η e είναι πολύ περίπλοκη. Στη χώρα προέλευσης του αιτήματο. η διαδικασία είναι περίπλοκη. Υπάρχουν πολύ σύντομες προθεσμίες για αυτά τα θέματα. Το έντυπο είναι πολύγλωσσο και δεν υπάρχει κανένας πραγματικό έλεγχος δεδομένη της περιπλοκότητας των ανταλλαγών ανάμεσα σε αρμόδιες αρχές. Δεν υπάρχει κανένα δε χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή για τους τομείς αυτού που καλύπτει η οδηγία. Ο τομέας ο είναι ο, αυτός που ενδιαφέρεται περισσότερο για αυτή την οδηγία, αλλά και είναι και ο τομέας που ε, υπάρχουν τα περισσότερα προβλήματα. Όπως μας θύμισε και η κυρία Εύελιν Γκέμπχαρντ, ε, ούτε στα θέματα ασφάλισης δεν είναι, ισχύουν τα ίδια πράγματα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει να λυθεί και να προσθέσω κάτι ακόμα, πολύ γνωστό, στη, στη Γαλλία τουλάχιστον, δεν ξέρω αλλού, αλλά στη Γαλλία δεν υπάρχει κανένα κεντρικό φάκελος όσον αφορά τις πτωχεύσεις, ε, τις δικαστικές ε, εκαθαρίσεις κτλ. Μπορεί δηλαδή κανείς να είναι υπό πτώχευση σε ένα νομό και στον άλλον να στήσει καινούργια επιχείρηση. Και την... Μπορεί μια εταιρεία να κάνει κάτι τέτοιο λοιπόν σε άλλη χώρα, χωρίς καμία προστασία για τον καταναλωτή ούτε για τους μικρούς πιστωτές. Τα πρακτικά προβλήματα λοιπόν εδώ δεν εξετάστηκαν πιστεύω σε αυτό, στη σύνταξη αυτού του κειμένου και εγώ συμφωνώ με την και, ε, τη συγγήτρια για την ώρα το EFTD είναι υπέρ της απόρριψης αυτής της πρότασης. Σας ευχαριστώ. Thank you Ευχαριστώ. Αν δεν θέλει κανένας άλλος βουλευτής το λόγο θα ήθελα να ε, δώσω το λόγο στην Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. να απαντήσω στο πρώτο σχόλιο της κυρίας Γκέπχαρτ. Νομίζω ότι υπάρχει μια παρανόηση. Αυτό που είπε η Κομισιόν είναι ότι το κείμενο δεν είναι τέλειο και σας καλέσαμε αυτόν τον τρόπο να το βελτιώσετε. Ε, όχι ότι είναι για τα σκουπίδια, δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις του κ. Μπούντα και της κ. Γκέπχαρτ. Ε, υποβλήθηκαν γραπτός κατά τη διάρκεια της συνάντησης των σκιωδών. Περιμέναμε και σήμερα για να στείλουμε απαντήσεις, γιατί, φανταζό, γιατί νομίζαμε ότι ε, η προθεσμία υποβολής ερωτήσεων έλγε σήμερα το μεσημέρι στις 12. Οπότε είπαμε να περιμένουμε προκειμένου να απαντήσουμε συνολικά σε όλες αυτές τις ερωτήσεις. Μόλις Φτάνουν στα χέρια μας οποιασδήποτε πρόσθετες ερωτήσεις έχουν τεθεί τον τελευταίο καιρό από την συνάντηση των σκιωδών και μετά, τότε θα στείλουμε για τις απαντήσεις. Οι πρώτες απαντήσεις είναι ήδη έτοιμες. Απλά ε, περιμένουμε τις πρόσθετες ενδεχομένω ερωτήσεις που θα έχουν φτάσει τον τελευταίο καιρό. Οπότε αν δεν υπάρχουν πρόσθετες ερωτήσεις, οι απαντήσεις θα σταλούν σήμερα ήδη το βράδυ. Αν έχουμε και άλλες βέβαια ερωτήσεις θα περιμένετε λίγο ακόμα. Υπάρχουν πολλές και διάφορες γνώμες σε αυτή την Επιτροπή για, το, για την αξία της ηλεκτρονικής κάρτας. Η ηλεκτρονική κάρτα είναι πράγματι ένα από τα εργαλεία που βοηθούν τους ε, ε, παρέχοντες υπηρεσίες. Ε, έχουμε το πόρταλ, έχουμε ε, την, ε, σε και κλπ. Η ηλεκτρονική κάρτα όμως ε, συμπληρώνει όλα αυτά. Ε, πρόκειται για ένα εργαλείο πρόσβασης αγορές, όχι για εργαλείο ενημέρωσης. μικροί συνήθως παρέχοντες υπηρεσίες μπορούν μέσω της ηλεκτρονικής κάρτας να βρουν το δρόμο τους μέσα στην γραφειοκρατία η οποία πολλές φορές τους βαραίνει και μάλιστα στην γλώσσα τους. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά να πω ότι η ηλεκτρονική κάρτα βοηθάει. Δεν είναι μαϊκή ράβδος. Και πάλι θα εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια και φραγμοί. Όμως, νομίζω ότι με αυτή την ηλεκτρονική κάρτα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι μικροί σχετικά παρέχοντες υπηρεσίες θα διευκολυνθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκέπχαρτ θέλει να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, και ευχαριστώ και τον ε, κύριο Μπούντα. Ε, παρότι έχουμε διαφορετικές απόψεις, θέλω να ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε αποτελεσματικά και να διορθώσω δύο πράγματα σε αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρώτον, ε, είναι αλήθεια το ότι αυτό αυτά που είπε η Επιτροπή δεν τα είπε την τελευταία εβδομάδα στο Στρασβούργο, αλλά σε μια δημόσια ε, εκδήλωση στις Βρυξέλλες την προηγούμενη εβδομάδα και εκεί εγώ ε, είπα κατά λέξη τι είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι το κείμενο δεν είναι καλό ότι δεν έχει διατυπωθεί σωστά. Και νομίζω ότι αυτό δεν το λέει ο κάθε υπάλληλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για το κείμενό του. Γι' αυτό με εντυπωσίαση. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχει εκπνεύσει καμία προθεσμία. Εγώ τις ερωτήσεις τις είχα καταθέσει στους ε, σκιοδησηγητές πριν από τη συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουν να προσθέσουν επιπρόσθετες ερωτήσεις. Και την προηγούμενη εβδομάδα παρακαλέσαμε την Επιτροπή να απαντήσει το συντομότερο δυνατόν. Θα ήθελα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τηρεί όλα αυτά που συμφωνούμε και να μην ε, λέει ιστορίες και ψέματα για το τι συνέβη και το τι δεν συνέβη. Με πάση περιπτώσει, ελπίζω να δοθούν πλέον οι απαντήσεις σε όλα αυτά τα δικά μας ερωτήματα γιατί πράγματι ο τρόπος ε, με τον οποίο η Επιτροπή ε, μεταχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι επιλήψιμος. Και θέλω για άλλη μια φορά να καταστήσω σαφές ότι Εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα να έχουμε μια εύρυθμα λειτουργούσα κοινή αγορά και με ενδιαφέρει η ελευθερία στην παροχή υπηρεσιών και στην επιχειρηματικότητα. Οι ελευθερίες αυτές να είναι υψηλού επίπεδου, καλής ποιότητας, αλλά ξέρετε να πω και κάτι άλλο. Για τη δική μου την πολιτική ομάδα αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι σε υψηλό επίπεδο όσον αφορά το εργασιακό δίκαιο, την προστασία του καταναλωτή και την κοινωνική κοινωνικής συνοχής στα κράτη-μέλη. Ειδικά λοιπόν σε περίοδους όπως είναι η σημερινή, όπου πολλοί πολίτες είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ως προς τα μηνύματα που εκπέμπουμε προς τα έξω. Ε, κατά πόσον δηλαδή δεχόμεθα κάτι χωρίς κανόνες ή κατά πόσον λέμε με απόλυτη σαφήνεια ότι θέλουμε άνοιγμα των αγορών αλλά σε υψηλό επίπεδο. Εσείς κύριε Μπούντα ε, αναφερθήκα στους αρχιτέκτονες. Οι αρχιτέκτονες δουλεύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αρχιτέκτονες δεν χρειάζονται επιπρόσθετα εργαλεία. Έχουν την οδηγία περί παροχής υπηρεσιών που τους καλύπτει, έχουν τους απαραίτητους φορείς. Εγώ ξέρετε έχω μιλήσει με αρχιτέκτονες και ε, όσον αφορά άλλα επαγγέλματα ε, τα οποία ε, καλύπτονται υποτίθεται από την τη νέα οδηγία μίλησα μαζί τους και μου είπαν ότι και αυτοί είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι με όσα ισχύουν μέχρι τώρα τις πληροφορίες που χρειάζονται για τη συνεργασία των διοικήσεων τις έχουν ήδη σας λέω εγώ ακούω τι έχουν να πούν οι επαγγελματίες, οι άνθρωποι της αγοράς και αυτοί μου λένε αυτά που προτείνετε τώρα είναι παντελώς περιτά. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ επιμένω δεν είμαι πεπισμένη ότι αυτό είναι ένα εργαλείο που χρειαζόμαστε. Εφόσον υπάρχουν άλλα εργαλεία, και εντάξει γνωρίζω ότι κάποια εργαλεία υπολείπονται, δεν είναι τέλεια, ε, καλύτερα να βελτιώσουμε αυτά που υπολείπονται για να λειτουργούν καλύτερα και όχι να προσθέσουμε άλλο ένα εργαλείο στην αγορά και κάποια στιγμή οι επαγγελματίες και οι επιχειρηματίες δεν θα γνωρίζουν ποιος είναι αρμόδιος γιατί. Δεν νομίζω ότι αυτό βοηθάει βοηθάει στην επιχειρηματικότητα. Ο κ. Μπούντα, εν συντομία παρακαλώ. Μάλιστα, Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομο. Δεν συμφωνώ με τα όσα είπε η Κομισιόν, γιατί η προθεσμία αφορούσε και τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Εν πάση περιπτώσει, τώρα υπάρχουν αρκετά μέσα και εργαλεία στην αγορά η Κομισιόν θα πρέπει να υποβάλει προτάσεις για εργαλεία που αφορούν κατηγορίες που δεν έχουν άλλα ή επαρκή άλλα εργαλεία. Μπορεί να υπάρχουν κάποια εργαλεία. Αυτή η ηλεκτρονική κάρτα όμως συμπληρώνει τα όσα υπάρχουν. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, η προθεσμία για τροπολογίες είναι η 1η Δεκεμβρίου αν δεν πλανώμε. Οπότε κλείνουμε αυτό το θέμα και περνάμε στο επόμενο και κλεισμένο των θυρών. Οπότε όποιος δεν έχει δικαίωμα να παρίσταται παρακαλώ πολύ να εγκαταλείψει την αίθουσα.